Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφοι, πριν από δύο εβδομάδες ήμουν στη Βέστερ Πλατ στον εορτασμό της ε, περτίου, ε, από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που θέρισε πολλά θύματα, εκατομμύρια θύματα στην Ευρώπη. Δεν θα πρέπει ουδέποτε να ξεχνούμε ότι η βία και ο πόλεμος μπορούν κάποια στιγμή να επανέλθουν στην Ευρώπη. Ε, γιατί τότε συνέβησαν και διάφορες άλλες ε, ε, βίαιες ενέργειες. Δύο υπάλληλοι της πολιτοφυλακής της Ισπανίας δολοφονήθηκαν από την ΕΤΑ εν υπηρεσία. Με μεγάλη θλίψη επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω για το θάνατο πρώην Βέλγου Ευρωβουλευτή του κύριου Έρνεστ Γκλίν που απεβίωσε στις 10 Αυγούστου σε ηλικία 78 ετών. Ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 1968 ε, μέχρι το 1994. Με ιδιαίτερη λοιπόν θλίψη θα ήθελα να σας ενημερώσω και για, την, ε, για το θάνατο ενός πρώην Βρετανού Ευρωβουλευτή, του Σερ Κρίστοφερ Πράουτ απεβίωσε στις 12 Ιουλίου σε ηλικία 67 ετών. Ο Σερ Κρίστοφερ, αργότερα Λόρδος Κίνξλεντ, ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 1990 μέχρι το 1994 και ήταν και πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών το 1994. Πριν ξεκινήσουμε τις εργασίες μας, θα ήθελα να σας ζητήσω να κρατήσουμε ενός λεπτού συγγύη για δύο πρώην συναδέλφους που έδωσαν και αυτή τη μάχη τους ε, για την Ευρώπη που έφτασε σε αυτή τη σημερινή μορφή. Τα πρακτικά της συνεδρίας της 16ης Ιουλίου του 2009 έχει διανεμηθεί. Τα έχετε λάβει και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχουν παρατηρήσεις για τα πρακτικά αυτά. Δεν βλέπω να υπάρχουν παρατηρήσεις, οπότε τα πρακτικά εγκρίνονται. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έλαβα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα Συγγνώμη, μια άλλη πληροφορία θα ήθελα να σας δώσω πρώτα. Οι βελγικές αρχές ε, με ενημέρωσαν για την ανάκληση του κυρίου Ζαν Κλοντ Μπάλκο σε μια θέση που είναι συμβίβαστη με τη θέση του Ευρωβουλευτή με βάση το άρθρο 7 ε, της ε, πράξης για τη.